Poštovane kolegice i Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε ώστε να ξεκινήσουμε με την απογευματινή μας σημερινή συνεδρίαση. Θα έχουμε μια κοινή ακριβώς ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Κώστα, να την, να την χαιρετήσω την κυρία Κώστα, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού, καθώς επίσης και τους άλλους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας που προσήλθαν στη δική μας συνεδρίαση, στη δική μας αυτή συνεδρίαση, σε μια κοινή συνεδρίαση. Θα ανταλλάξουμε απόψεις ε, για την πολιτισμική διπλωματία σαν παρακολούθηση της δράσης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των δραστηριοτήτων της και θα ήθελα σε αυτό το σημείο δύο πραγματογνώμονες να χαιρετήσω την κυρία Ντάνα Ουστάτη που είναι διευθύντρια της More Europe όσον αφορά τις πολιτισμικές σχέσεις και τον κύριο Γκότφριντ Βάγνερ, σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πολιτισμικών θεσμικών οργάνων που ε, εργάζεται για την ΑΕΔΕΠ Καλώς ορίσατε λοιπόν και οι δύο. Οι σκέψεις μας για το πόσα οι. Ε, πολιτική μας, την πολιτισμική διπλωματία θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να ενδυναμωθεί και πώς μπορεί να διαμεσολαβήσει, να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο σε συγκρούσεις και σειράξεις είναι μια πρωτοβουλία που κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία από την ε, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είχε αναλυθεί. Προτού δώσω τον λόγο στους πραγματογνώμονες θα ήθελα στην κυρία Κώστα να δώσω τον λόγο πρώτα, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, και να την παρακαλέσω να μας πει δύο λόγια σχετικά με αυτές τις, για αυτές τις διαφορετικές δραστηριότητες και μέτρα που έχουν ε, αναλυφθεί μέσα στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που εντάσσονται κυρίως μέσα στο πλαίσιο της πολιτισμικής διπλωματίας. Έχει τον λόγο κυρία Πρόεδρε Κώστα. I will speak in Italian if you allow me. Θα μιλήσω στα Ιταλικά, αν μου το επιτρέπετε. Απλά για να υπερασπίσουμε την πολυγλωσία και την πολιτισμική πολυμορφία. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Αντιπρόεδρο Πλένκοβιτς και τον ε, κύριο Μπρόκ, τον Πρόεδρο, για αυτή την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που διεξάγουμε από κοινού. Πριν λίγο καιρό έγινε μια ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό μέσω των δράσεων των επιτροπών μας το Ευρωκοινοβούλιο να δώσει περισσότερη σημασία στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρώπης που να βασίζονται στην πρόθεση του διαπολιτισμικού διαλόγου, του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στις εξωτερικές σχέσεις. Οι πολιτισμικές σχέσεις λοιπόν και η συνεργασία σε αυτό το τομέα και οι πολιτιστικές ανταλλαγές ε, αποτελούν δομικά στοιχεία. Ειδικότερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές για την Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, για τον κόσμο. Μπορούν να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική συνεργασία της Ευρώπης. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την πρόκληση ως Ευρωπαίοι, αλλά όχι μόνο την πρόκληση κινδύνων φονταμεταλλισμού, ριζοσπαστικοποίησης που πολλές φορές ε, χρησιμοποιούν συγγνώμη, την ε, πολιτισμική διαφορά για να καταπνίξουν ε, τη δημοκρατία, τις ελευθερίες με ιδευθείς τρομοκρατικές πράξεις. Η πολιτισμική, η πολιτιστική διπλωματία λοιπόν, ο πολιτιστικός διάλογος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό χαρτί οριζόντιο για την εξωτερική μα πολιτική. Πρέπει να ενισχύσουμε στο σύστημα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη διάσταση του πολιτισμού. Κάτι που μας έκανε εντύπωση πρόσφατα στην Ολομέλεια του Στρασβιούργου ήταν η ομόφωνη ψήφος του Κοινοβουλίου ε, για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ότι σήμερα συχνά σε κοντινές χώρες με τις δικές μας ε, κοντά στη Μεσόγειο γίνονται επιθέσεις συμβολικές κατά πολιτιστικών συμβόλων θρησκευτικών σαν η πολιτιστική κληρονομιά να μετατρεπόταν σε ένα όπλο όπλο για, για το μη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην Επιτροπή μας ε, αποφασίσαμε να μαχηθούμε και σε αυτό το μέτωπο μετά από αυτή την ψηφοφορία επί εκείνης της έκθεσης ε, για τα θεμελιώδη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου συμπεριλήφθηκε μια τροπολογία ώστε τέτοιες πράξεις να θεωρούνται έγκληματα κατά της ανθρωπότητας. Πιστεύω χρειάζεται και περαιτέρω δράση, συγκεκριμένες προτάσεις για να αναλάβουμε ευθύνε. Στην Επιτροπή Πολιτισμού, όπως υπενθυμίσατε, στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, εγκρίναμε το 2011 μια έκθεση για την πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτήν ζητάμε να ενταχθεί πιο εκτενώς ε, αυτός ο τομέας ε, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το ζητήσαμε και, στην ε, και από την ύπατη εκπρόσωπο κατά την παρουσία της εδώ στο Κοινοβούλιο. Τη ζητήσαμε να υπάρξει ισχυρότερη συνεργασία ώστε να αρχίσουμε να μιλάμε για μια πιο κοινή ε, πολιτική πολιτισμού συμπεριλαμβάνοντας τους στόχους, τους πολιτιστικούς διαλόγους, τον κοινωνικό διάλογο και την νέα νοοτροπία μιας νέας εταιρικής σχέσης, όχι μόνο με τη Μεσόγειο αλλά και με τις χώρες ε, που βρίσκονται ανατολικά της Ευρώπης, ώστε να είναι αισθητή αυτή η διάσταση και πρέπει πιστεύω να εργαστούμε πιο εντατικά για την προστασία, την πρόληψη και τη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς που υπενθυμίζω ανήκει σε όλους, όχι μόνο στις χώρες όπου βρίσκονται, όπου βρίσκεται η πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης τίθεται και το ζήτημα της ενίσχυσης του πολιτιστικού τομέα, του οπτικοακουστικού τομέα, των διαφόρων τρόπων έκφρασης του κινηματογράφου, να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για μια νέα ανταλλαγή ε, ανθρώπων, μέσων. Ζητείται συχνά από άλλες χώρες αυτό, να υπάρξουν ανταλλαγές πανεπιστημιακές, ε, πολιτισμικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών ιδρυμάτων, ώστε να δώσουμε όθηση σε όλα τα μέσα που υπάρχει, υπάρχουν σε αυτό το τομέα, σκέφτομαι τώρα το ψηφιακό τομέα, υπάρχουν δυνατότητες ε, κινητικότητας των καλλιτεχνών, των δημιουργών, των έργων. Πρόσφατα ως Κοινοβούλιο προσαρμόσαμε την οδηγία για την επιστροφή των κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών. Ε, είναι ένα θέμα που ακόμα παραμένει ανοιχτό. Θίξαμε και το θέμα της συνεργασίας για την γνώση και το σεβασμό των πολιτιστικών ταυτοτήτων και των πολιτιστικών μειονοτήτων. Πιστεύω ότι μπορούμε μαζί να κάνουμε κάποιες κινήσεις ε, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Και ήθελα επίσης να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία του κύριου Σούλτ με τον κύριο Ταγιάννη για το διαθρησκευτικό διάλογο, δύο διασκέψεις που θα λάβουν χώρα και όπου θα συνεργαστούμε με άλλους συναδέλφους, διότι είναι κάτι απαραίτητο. Χρειάζεται πρώτα να γνωρίσουμε πώς έχουν τα πράγματα πριν ξεκινήσουμε το διάλογο. Θεώρησα λοιπόν ότι σήμερα θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε αυτόν τον προβληματισμό για αυτές τις κοινέ πολιτικές ξεκινώντας από ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που είδαμε τα τελευταία χρόνια όπου η Επιτροπή Πολιτισμού υποστήριξε την προπαρασκευαστική δράση που ονομάζεται More Culture from Europe and the World και που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια από οκτώ ε, πολιτιστικούς οργανισμούς σε συνεργασία με το δίκτυο EUNIC με τη συμμετοχή 16 γειτονικών χωρών και 10 στρατηγικών εταίρων. Προσιαστώ στον Ιούνιο του 2014 τελική έκθεση. Οι εκλογέ, η νέα θητεία και η εκκίνηση των εργασιών μα δεν μα επέτρεψαν να το συζητήσουμε πρωτήτερα. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα που δεχτήκατε αυτή την πρόταση εδώ στην Επιτροπή ΑΦΕΤ να δούμε μαζί τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν από αυτό το πείραμα, να προβληματιστούμε επί αυτών, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, από μια αφετηρία πιο ε, σταθερή από απλές ε, κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά είχα να πω και θα δώσω τώρα το λόγο, εγώ ή εσείς δεν ξέρω, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου αλλά που περιλαμβάνουν και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που πιστεύω θα ενδιαφέρουν και εσά. Καλό είναι λοιπόν να συζητήσουμε. Δίνω το λόγο λοιπόν, αν μου το επιτρέπετε, κύριε Βλέγκοβιτ, στην Σάνα Ουστάτη, διευθύντρια τη More Europe External Cultural Relations και στον Gottfried Wagner, σύμβουλο έργων για την πρωτοβουλία More Europe για τα Ιδρύματα Πολιτών και τα Πολιτικά Ιδρύματα για τον πολιτισμό στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις. Θα μιλήσουμε φαντάζομαι με τη σειρά με την οποία αναφέραμε προηγουμένω, κύριε Οστάτη. Έχετε δέκα λεπτά. Δέκα λεπτά ο καθένα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτέ, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα εκ μέρους του Κοσότιου που έχει ετοιμάσει την ε, δοκιμή το πείραμα αυτό όσον αφορά τις εξωτερικές πολιτισμικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στο κοσόρτιουμα αυτό και όσους συνεργάστηκαν με την ε, θέση σε εφαρμογή των ιδεών αυτών. Σας ευχαριστώ επίσης που μου δώσατε την ευκαιρία σε αυτήν την ε, κοινή συνεδρίασή σας να έρθω να σας μιλήσω για την ε, πολιτισμική διπλωματία και για τις προπαρασκευαστικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Πολιτιστικής Επιτροπής, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών που βρίσκονται εδώ σήμερα. Η πολιτισμική Διπλωματία λοιπόν και εξωτερικές σχέσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που δεν αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδίου. Είναι ε, σημαντικά στοιχεία για τις χώρες μέλη, για την ε, Ευρώπη, για τους καλλιτέχνες, για τους πολιτιστικούς παράγοντες, αλλά και για την κοινωνία των πολιτών τόσο της Ευρώπης όσο και άλλων τρίτων χωρών είτε που γειτονεύουν μαζί μας, είτε που συμμετέχουν σε κοινέ δράσεις μαζί μας. Τι έχουμε διαπιστώσει μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεις και έρευνες. Προηγουμένως όμως επιτρέψτε μου δύο-τρία λεπτά να σας εξηγήσω ποιο είναι το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανακοινωθεί η προπαρασκευαστική μας δράση. Όπως ήδη είπε η κυρία Σίλβια Κώστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα όσον αφορά τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που τονίστηκαν αυτά στην Επιτροπή Πολιτισμού περιλαμβάνουν διάφορα σημαντικά στοιχεία και έχω να προσθέσω και εγώ μερικά παραπάνω από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας δώσω μια πλήρη εικόνα του γενικού πλαισίου. Πρώτα απ' όλα τι λέει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 167 παράγραφος 3 που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη να προωθήσουν τις πολιτιστικές επιτυχίες στις διεθνείς σχέσεις. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μέρος μιας σύμβασης του 2005 της UNESCO δηλαδή όσον αφορά την πολιτισμική πολυμορφία και βάσει αυτής της σύμβασης έχει την υποχρέωση την πολιτιστική διάσταση να την κάνει σημαντικό στοιχείο των εξωτερικών της σχέσεων. Ένα άλλο σημαντικό πλαίσιο που πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό και τον τρίτο πυλώνα που έχει ως στόχο να προωθήσει το ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στην υποσλοβενική Προεδρία και την έκθεση Σχράκερ επίσης και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ακολούθησαν διάφορες πολιτικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα και ποια είναι αυτά. Από το 2011 μέχρι το 2014 πολλές ευρωπαϊκές προεδρίες οργάνωσαν συναντήσεις με αξιωματούχους από διάφορα Υπουργεία Πολιτισμού ή Εξωτερικών Υποθέσεων. Από τις συναντήσεις αυτές είχαμε ένα νέο βήμα ανταλλαγής απόψεων στις εξωτερικές σχέσεις για πολιτισμικά θέματα με μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση ΙΑΚ ε, χρησιμοποίησε μία ομάδα για την πρόσθεση των ε, εξωτερικών σχέσεων μέσα από τη διάσταση του πολιτισμού και σαν ε, παράδειγμα πήραν την Κίνα. Ξεκίνησαν από την ιδέα ότι είναι μια προστιθόμενη, προστιθέμενη αξία ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις, άπαξ δηλαδή και διμερός υπάρχουν τέτοιες σχέσεις, να υπάρχουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2013 λοιπόν το Συμβούλιο ανέφερε προσδοκίες για συγκεκριμένες δράσεις που θα έπρεπε να αναλυθούν στις πολιτιστικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Να δοκιμαστούν δηλαδή σε αυτά τα πλαίσια κάποιες δράσεις και αργότερα να επεκταθούν και παρετέρω. Έτσι χαρτογραφήσαμε το τοπίο στις πολιτισμικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, που ήταν το πρώτο βήμα για διάφορες ευκαιρίες και προκλήσεις, αλλά και νέες ιδέες που θα μπορούσαμε να είχαμε στην πολιτισμική συνεργασία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες εξελίξεις που έλαβαν χώρα ήταν στην εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης, στο, σχετικό, δικό τους δηλαδή πολιτιστικό συμβούλιο, με υπηρεσίες για την ένταξη της πολιτιστικής διάστασης σε μέσα όπως είναι εκείνο της εταιρική ε, σχέσης ή της σταθερότητας και της ειρήνης. Το 2014 επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης οργάνωσε και ένα σεμινάριο για τον πολιτισμό σε χώρες όπου υπάρχει σύγκρουση για να δούνε τι συμβαίνει εάν λάβουμε υπόψη μας τον πολιτισμό σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν υπήρξαν συγκεκριμένες συστάσεις από τους συμμετέχοντες. Κάποιες από αυτές τις συστάσεις εφαρμόζονται στα πλαίσια του μέσου για την ειρήνη. Επιπλέον από τις εξελίξεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό για την προπαρασκευαστική δράση στις εξωτερικές σχέσεις που εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ενός consortium υπό του Ινστιτούτου More Europe σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Άμστερνταμ, με τις Μποζάρα στις Βρυξέλλες και άλλων οργανώσεων. Η CPDM, ένα acting, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Δανέζικο Πολιτισμικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Σχέσεων της Τουσγάρδης. Με έντονη συμμετοχή διαφόρων ε, διάσημων εμπειρογνωμόνων. Η προπαρασκευαστική δράση είχε σαν στόχο τον προβληματισμό και τις εξελίξεις προκειμένου να ισχυθεί ο ρόλος του πολιτισμού στις εξωτερικές ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα αυτό. Όπως είπαμε ήδη καλύπτονται 16 χώρες από τις γειτονικές, 10 ε, από τη στρατηγική εταιρική σχέση και υπόλοιπε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 26 επίσης ε, εκθέσεις για μεμονωμένες χώρες και συστάσεις για ε, δοκιμαστικά προγράμματα. Η προπαρασκευαστική δράση μας λέει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για τον πολιτισμό στις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνει ότι πάρα πολλοί στον κόσμο ενδιαφέρονται πάρα πολύ να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις από κοινού με την Ευρώπη. Πριν δώσω το λόγο στο Βίλφιντ Βάκνερ, επιτρέψτε μου να αναφέρω και δύο ακόμα συστάσεις που εμεί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικές. Πρώτον, οι πολιτιστικές σχέσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στην ε, παρουσίαση ε, ευρωπαϊκών πολιτιστικών ε, εκδηλώσεων προς τους άλλους. Όχι. Πρέπει να δείξουμε την πολυμορφία του πολιτισμού στην Ευρώπη, να βοηθήσουμε για την δημιουργία ικανοτήτων και να υπάρχει στενή συνεργασία. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην κυβερνητική ευθύνη και τις αυτόνομες πρακτικές στον τομέα της τέχνης. Και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση που μας αποστήλατε να συμμετάσχουμε σε συζήτηση σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή με τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Επέστρεψα από την την Ισία, όπου υπήρξε η επίθεση στο Μουσείο Μπαρδόμπου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξή μου και η απογνωσή μου για την επίθεση αυτή και για τις αξίες της δημοκρατίας και του πολιτισμού που υπέστησαν αυτό το πλήγμα. Η συνάντησή μας εδώ λοιπόν γίνεται σε μια κατεπίγουσα χρονική στιγμή κατεπηγόντως ε, είναι ανάγκη να αντιδράσουμε. Και όχι μόνο με το να αναφέρουμε τις συστάσεις για τις δράσεις και έχετε και τα έγγραφα, αλλά θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα προτείνουμε κάποια θέματα που πρέπει να τεθούν υπό συζήτηση. Πρώτα απ' όλα το κύριο αποτέλεσμα της ε, δράσεις μας είναι τα τεκμήρια. Υπάρχουν τεκμήρια ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό για τον πολιτισμό ως τμήμα και μέρος της εξωτερικής πολιτικής δράσης πέρα από τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Είναι ένα δυναμικό για ευρωπαϊκή δράση συνολικά. Υπάρχει και εκπληκτική ζήτηση και αυτό το καταδεικνύουν όλες οι μελέτες και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τα κράτη-μέλη που έχουν κατανοήσει ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον η Ευρώπη η ίδια να αναλάβει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πολιτισμικά τρίτων. Το ανέφερε η κυρία Οστάτη. Υπάρχει ευρύτατη βάση συμφωνίας. Όταν κάνουμε λόγο για την πολιτισμική διπλωματία σήμερα υπάρχει μια νέα έννοια για αυτήν. Αφού γραζόμαστε ακούμε βασιζόμαστε στην αμοιβαιότητα, στον σεβασμό αμοιβαία. Είναι λοιπόν μια συνεργασία αμοιβαία. Και τέταρτον, μην ξεχνάμε τη δραστηριοποίησή μας σε ένα περιβάλλον εντονότατου ανταγωνισμού. Καλού αλλά και λιγότερο καλού ανταγωνισμού. Και η Ευρώπη πρέπει λοιπόν εδώ να δράσει αποτελεσματικά. Το οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους ε, στις προπαρασκευαστικές δράσεις ε, τόνισαν ότι στο τέλος τέλος θα είναι μια κατάσταση κέρδους win-win για όλους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και τα κράτη-μέλη και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο καινοτόμο στοιχείο δεν είναι ο ένας εναντίον του άλλου είναι μια αμοιβαία δράση που εμπλουτίζει αμφωτέρωθεν να μην ξεχνάμε και την κοινωνία των πολιτών που τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να υπάρχει μια διακρατική, μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα πολιτισμική τέτοια πρωτοβουλία. Είναι επίσης win-win, κέρδους, κατάσταση, τελικού ωφέλους όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση. Κάνουμε λόγο για την ε, συνάθρηση, το άθροισμα του δυναμικού μέσω των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών σε αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχει η βούληση να δούμε την δυνατότητα να προσθέσουμε, να αθροίσουμε δυναμικό και ώστε να διευρυνθεί αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ακριβώς που χρειαζόμαστε. Και η κύρια έννοια όταν κάνουμε λόγο για τις μελλοντικές ε, ε, εναλλακτικές στρατηγικές δυνατότητες είναι η αλληλοσυμπληρωματικότητα, η παραπληρωματικότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τα επόμενα βήματα. Βήματα που θα στοχεύουν και θα προσανατολίζονται με ε, δράσεις πολιτικές και πολιτισμικές. Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο για να προωθηθεί αυτού του είδους ε, ή στρατηγικού χαρακτήρα δράση. Αναμένουμε, αναμένουν όλοι μετά από τόσα χρόνια, τώρα τις, μετά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, την πραγματική ουσιαστική δράση που θα οδηγήσει σε πραγματικά αυθεντικά αποτελέσματα. Να αναφέρω κάποιες ε, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που βρίσκονται υπό εξέλιξη οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν μια συνολική εικόνα του τι συμβαίνει. Έχουμε για παράδειγμα μια νέα, ένα νέο πρόγραμμα πολιτικής γειτονίας ε, σε σχέση για παράδειγμα με το ίδιο το Κίεβο ξεκινώντας ε, την δημιουργία δυναμικού και οικοδόμησης ε, αμοιβαία δράσης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα για παράδειγμα όσον αφορά την, Ισία που αναφέρεται και από πλευράς της αντιπροσωπείας σχέσεις αδερφοποίησης μεταξύ Αζερβαϊτζάν και κρατών μελών να υπάρξει μεταρρύθμιση της πολιτισμικής πολιτικής ε, σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Έχουμε και τον ορίζοντα 2020 για το, την έρευνα, για την ε, πολιτισμική δράση και επιστημονική δράση μέσα σε ένα πλαίσιο επιστημονικών πρωτοβουλειών για την πολιτισμική διπλωματία της Ευρώπης. Να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητά μας από πλευρά μας και υπάρχει μεγάλη αναζωογόνηση, νέο δυναμικό σε σχέση με αυτές τις δράσεις από πλευράς μας. Η κυρία Στάτη ανέφερε κάποιες πρακτικές ε, δυνατότητες που προετοιμάζονται. Το αμέσα και τα εργαλεία για την εξωτερική πολιτική αφενός εργαλεία και μέσα που συνεισφέρουν για τη δημιουργία σταθεροποίησης και σταθερότητας. Θα, ήδη από το, το 2016 θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα ως δυνατότητα. Θα έχουμε νέα φεστιβάλ ταινιών και κινηματογράφου και σε τρίτες χώρες. Ένα δίκτυο δημιουργών, νέων δημιουργών. Διευκολύνεται αυτό και από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτό. Σταυροδρόμια πολιτισμού, δίκτυα με, με κρατικά πολιτισμικά όργανα και φορείς και κατανοώ και γνωρίζω ότι υπάρχουν νέες δυνάμεις για να ενδυναμωθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και στο εξωτερικό πεδίο όσον αφορά τις πολιτισμικές δράσεις στο πεδίο του πολιτισμού και της παιδείας. Και η ενημέρωση και πληροφόρηση δίνει πολλές δυνατότητες. Αυτό το φθινόπωρο θα έχουμε ένα πολιτισμικό φόρουμ ως ε, πρωτοβουλία. Θα μαζευτούν εκατοντάδες ε, εμπλεκόμενοι από όλη την Ευρώπη και ελπίζουμε φυσικά και ότι η κυρία Μογκερίνη, είπατε εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμμετάσχει. Πού θα κατευθυνθούμε τελικά δεν το γνωρίζουμε ε, κάποια χρόνια πριν είχαμε αυτή την ανακοίνωση που ε, δημιούργησε ε, στην ημερήσια διάταξη στο θεματολόγιο για τον πολιτισμό και τις πολιτισμικές δράσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα είναι πραγματικά αξιόπιστο και αποτελεσματικό. Πού χρειάζονται τέτοιες δράσεις τώρα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω πέντε κύρια πεδία χωρίς να επισέλθω υπερβολικά σε λεπτομέρειες. Πρώτα και κύρια θα έλεγα αυτό που χρειαζόμαστε είναι δράση όσον αφορά συγκρούσεις και σειράξεις και πρωτοβουλίες πολιτισμικές, πολιτισμικής, πολιτισμικής διπλωματίας. Όχι μόνο μεταξύ α, κρατών της Ανατολής και του Νότου, αλλά και τρίτων χωρών. Και το δυναμικό το οποίο εδώ αφορά και την κατάρτιση και την παιδεία και την εξειδίκευση. Τρίτον, και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το αρχικό πλαίσιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες, δυσχερείς καταστάσεις και να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα και τα θέματα του Ιράν. Η συμφωνία για τα θέματα εκμετάλλευσης ε, ατομικής ενέργειας από πλευράς του Ιράν και να δούμε πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλίες να συνεισφέρει. Οι νέοι Ιρανοί πραγματικά αναμένουν να πάνε Ευρωπαίοι στη χώρα τους, στο Ιράν και να συνεργαστούν μαζί τους σε αυτούς τους τομείς. Τέταρτον, κοινωνία των πολιτών. Η ε, πολιτισμική δράση έχει κύρια, κυριότατο χαρακτήρα να υποστηρίξει τις ε, αλλαγές και την καινοτομία. Και πέμπτο, οι επαφές ε, για την προώθηση των πολιτισμικών σχέσεων. Για να σημειωθούν πρόοδοι σε αυτά τα πέντε πεδία χρειαζόμαστε κάποια τεκμήρια και αποδείξεις ότι διαχειριστικά μπορούμε να πετύχουμε κάτι συναθρίζοντας και προσθέτοντας δυναμικό. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού λοιπόν θα ε, αναμένουν το να μπορέσουν να ε, ε, αναλυφθούν τέτοιες δράσεις χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω επιβαρύνσεις ή δυσκολίες. Δυσ, δυνατότητες να συναθρήσουμε, να προσθέσουμε δυναμικό, να διευρύνουμε δυνατότητες και να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, να βρούμε νέους τύπους και μορφές πως μικρές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συνεργαστούν σε ένα δεδομένο πλαίσιο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεύτερο, χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε επίσης νέες μεθόδους ώστε να προσθέτουμε και να εξεύρουμε νέο δυναμικό και νέους πόρους ε, ώστε να υπάρχει εταιρική ευθύνη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διότι κατανοούν την ανάγκη να υπάρξει πολιτισμική επικοινωνία και εδώ πρέπει ακριβώς η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων να αναπτυχθεί να μπορέσουν να υποστηριχθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε σχέση με άλλες χώρες. Και τρίτον, ο ευδιάκριτος χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της Ευρώπης, με α, οπωσδήποτε νέες ευφυείς μεθόδους χρήσης νέων τεχνολογιών, ώστε να υπάρξει απήχηση αυτής της ευρωπαϊκής πολιτισμικής διπλωματίας σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Τε, τελευταίο στοιχείο, πώς μπορούν οι δύο κοινοβουλευτικές μας επιτροπές να δράσουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν στα όσα βρίσκονται υπό εξέλιξη στο pipeline για την, εξωτερική, ε, για την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Εδώ πρέπει δύο στοιχεία, δύο άξονες να δούμε, δύο εκκλήσεις που απευθύνονται από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και από ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις από την Αυστρία. Ζητείτε να βοηθηθούν από τα θεσμικά όργανα, να υπάρξει το αναγκαίο σωστό θεσμικό πλαίσιο. Χρειάζονται διευρυμένες πολιτικές για τους προσανατολισμούς για να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία που πρέπει να υπάρξει. Για το ποια μέσα και ποια εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δεν είναι δική μου δουλειά να το καθορίσω αυτό, αλλά πρέπει οι νέες αυτές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της, πολιτικής, Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, να μπορέσει να δώσει τους σπόρους να αναπτυχθεί μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και τρόπο αυτό το πλαίσιο για τη στρατηγική σημασία πολιτισμική αυτή δραστηριοποίηση. Και επανέρχομαι τώρα στο ε, ε, σημείο για τη δράση όχι μόνο χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ε, σχεδιασμό και προγραμματισμό που έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα αλλά και βραχυπρόθεσμα άμεσα πρέπει να είμαστε δυνα... ικανοί να δράσουμε άμεσα και να δραστηριοποιηθούμε. Γιατί να μην έχουμε μία μονάδα άμεσης αντίδρασης και δράσης πολιτισμικά που θα βοηθά τους ανθρώπους επιτόπου. Για παράδειγμα, για το εικονικό μουσείο της Μοσούλης, για τα όσα καταστράφηκαν από τον πολιτισμό, από την οίκης ώστε να μπορούν, για παράδειγμα, σε σχέση με το Κίεβο, μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών να υπάρχουν τέτοιε επαφέ. Θα μπορούσα πολλά παραδείγματα να δώσω. Αυτά που χρειάζονται είναι τα κονδύλια, οι δυνατότητε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα άτομα, να συνεχίσουν τι πρωτοβουλίε και τι δράσει του, ώστε να προχωρήσουμε. Είναι ένα θέμα ο σχεδιασμό, προγραμματισμό, μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά είναι εξίσου σπουδαίο ζήτημα το να υπάρχει μια μονάδα άμεση δραστηριοποίηση και δράση, ώστε να μπορούμε άμεσα να αντιδράσουμε στις ανάγκες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Βάγνερ. Ας ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτησή μας. Ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο είναι ο κύριος Μιλανών. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κώστα πρόεδρο τη Επιτροπής Πολιτισμού αλλά και τον κύριο Μπροκ που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη συνάντηση αυτή. Ο πολιτισμός πιστεύω ότι ήταν ε, πάντα ένας πολύ καλός σύμμαχος της διπλωματίας με κοινέ πολιτιστικές δράσεις που πάντα συνόδευαν τις καλές σχέσεις μεταξύ χωρών και λών. Εννοείται ότι αυτή η ήπια δύναμη, σύμφωνα με τον Τζόσεφ Νάιν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε και εμείς ότι είναι κάτι που βοηθάει. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης, το είπε και η κυρία Κώσταλο και ο κύριος Βάγκνερ, πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός ε, κυρίως στη Μεσόγειο. Θυμόμαστε και την, ε, την Ισία τώρα. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να επιμείνουμε στην προσέγγιση των αξιών μας. Έχουμε συχνά κοινέ ρίζες. Άλλοι θέλουν να δουν ε, αντιφάσεις, συγκρούσεις πολιτισμών μερικές φορές. Εμείς λοιπόν θέλουμε να επιμείνουμε αντίθετα ότι οι δράσεις πολιτισμικές σε αυτές τις χώρες, διάλογος, ε, σεβασμός της πολυμορφίας είναι πράγματα που χρειάζονται. Και μην ξεχνάμε ότι πολύ πρόσφατα έχουμε μια κοινή ιστορία πολύ από εμά και περάσαμε από διάφορα στάδια φιλίας και πολιτισμικών ανταλλαγών. Ο πολιτισμός λοιπόν είναι ένας παράγοντας που μας θυμίζει και τις κοινέ μας ρίζες αλλά και τις κοινέ μας αξίες. Την ανοχή, την ποικιλομορφία, Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε ενισχύει την πολιτισμική παρουσία της Ευρώπης είναι κάτι θετικό και είναι κάτι που χρειάζεται. Ενώ πολλοί προσπαθούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια νοοτροπία διαλόγου και ανταλλαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μιλανόν, Τώρα το λόγο κύριος Λέρτς, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ θερμά, λέει ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ θερμά κυρία Κώστα για την πάρα πολύ καλή αυτή σύγκληση και ε, συμμετοχή των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών καθώς επίσης και για τα όσα είπατε που με ικανοποιούν είχα την ικανοποίηση και τη χαρά πριν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να έχω εργαστεί στο Ινστιτούτο Γκέτε και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η πολιτισμική συνεργασία και οι προσπάθειες και πρωτοβουλίες στον πολιτισμικό τομέα. Οι πρωτοβουλίες που και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλήφθηκαν ήταν στο επίπεδο του πολιτισμού μία ας το πω έτσι ομάδα διακομματική intergroup που δημιουργήθηκε για το θέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και τον τουρισμό ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, δηλαδή και συμβολική σημασία ότι κοινοβουλευτικοί πρόσωποι από διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές συμμετέχουν σε μια δυνατότητα διαλόγου, ώστε να αποσαφινιστούν τα θέματα της ε, θρησκευτική ιστορίας, αλλά και των πολιτισμικών θεμάτων. Δηλαδή, να δούμε ποιες είναι οι ρίζες μας, προερχόμαστε από την, ε, την δυνατότητα εκείνη που ε, στις ρίζες μας και στο σύμβολο το οποίο μας χαρακτηρίζει και τη γλώσσα και τα χαρακτηριστικά τα οποία ενδυναμώνουν τον πολιτισμό και τις γλώσσες μας διαδραματίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο Intergroup αυτό ε, μπορούν να ληφθούν υπόψη και να καλυφθούν αυτά, αλλά και πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που μπορεί να ε, προέρχονται και από μια ομάδα, για παράδειγμα, που πανευρωπαϊκά μπορεί να δράσει και που με βάση αυτές τις ε, δυνατότητες θα δημιουργηθεί μια κοινή δραστηριοποίηση που θα παρακολουθεί αυτές τις δράσεις ε, και που μπορούν να προσκληθούν ε, άτομα σε αυτή τη δυνατότητα που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο. Ένα άλλο περαιτέρω θέμα για το οποίο η, πολιτική, ε, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι το θέμα του 2018 που θα επικεντρωθούμε στο θέμα της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς. Να δώσουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό το θέμα και από κοινού να δράσουμε ώστε η ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά να μπορέσει να ενδυναμωθεί εσωτερικά, η ευρωπαϊκή ταυτότητα να ενδυναμωθεί όσον αφορά και την πολιτική γειτονία που αναπτύσσουμε και τις σχέσεις μας με άλλες ε, χώρες και άλλους λαούς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όλοι οι συναδελφοί να μην υπερβούν τα δύο λεπτά γιατί είμαστε πολλοί και οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν στις 6.30. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Διακόνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πραγματικά πολύ πρέπει να πω για το ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ και συζητούμε για αυτό το θέμα. Και να ρωτήσω και να πω γιατί, να το υπενθυμίσω το γιατί. Στη δεκαετία του 70, πριν από πολλά πολλά χρόνια, υπήρξε μία ομάδα, εγώ προέρχομαι από τη Ρουμανία και αυτή η θεατρική ομάδα, αυτός ο Θίασος ε, που μία φορά ε, είχε παρουσιαστεί και είχε συμμετάσχει στην πρεσβεία μας ε, στην Ουάσιγκτον. Εκείνοι που εργαζόντουσαν στην πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον ήρθαν σε εμάς τους ηθοποιούς και μας είπαν δεν μπορείτε να φανταστείτε κυρίες και κύριοι πόσο σημαντικά άτομα προσήλθαν σε εμά σήμερα σε αυτή την εκδήλωση που ποτέ δεν είχαν επισκεφθεί την πρεσβεία μας και που ποτέ δεν είχαμε επαφές μαζί τους. Ήρθαν τώρα με αφορμή αυτή τη θεατρική παράσταση που δώσατε εσείς στην πρεσβεία μας. Τότε κατανόησα πόσο σημαντική είναι η πολιτισμική διπλωματία ως δράση και με τους ε, διπλωμάτες που είχα έρθει σε επαφή τότε από τη χώρα μας για να ε, ε, δοθεί σάρκα και οστά και νέα ζωή σε αυτή την πρωτοβουλία θα ήθελα να πω ότι αυτή η έννοια φοβούμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ριζώσει και δεν υπάρχει στη Ρουμανία. Υπάρχουν πολύ πολλά θεσμικά όργανα πολιτισμικά που λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω χρειαζόμαστε αυτή την προσέγγιση, αυτή την έννοια που απουσιάζει ακόμα. Το ότι σήμερα συνεργαζόμαστε και βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε όλα αυτά τα θέματα εκφράζει την ελπίδα μου ότι μπορούμε να εκφράσουμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα ως κοινοβούλιο ότι οι χώρες μας, η χώρα μου για παράδειγμα θα έπρεπε να καταλάβουν και θα έπρεπε να καταλάβει και οι άλλες χώρες να αντιληφθούν ότι αυτό το μέσο είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματικό. Από τη ρωμαϊκή εποχή, από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μετά το στρατό χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι τον πολιτισμό. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν αυτός. Τρούπελ. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Τρούπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι Λυπάμαι που δεν παρευρίσκονται περισσότεροι συνάδελφοι. Θα ήθελα να εμπλακούν περισσότεροι εδώ συνάδελφοι από την ΚΑΛΤ και την ΑΦΕΤ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τη συμβολή τους. Θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι μόνο καλοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν για να ενταχθεί ο πολιτισμός ε, στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άμεση η ανάγκη, όπως βλέπουμε τώρα με τις διάφορες σειράξεις. Υπάρχει άμεση ανάγκη για διάλογο. Καλή είναι η διπλωματία από πάνω προς τα κάτω, αλλά πολλά μπορούν να επιτευχθούν με τη συμμετοχή των πολιτιστικών ιδρυμάτων, των NGO, της κοινωνίας των πολιτών και πολιτιστικών προγραμμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες. Η προσέγγιση αυτή προσθέτει αξία, διότι καθιστά δυνατή την προσέγγιση ανθρώπων που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να προσεγγίσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτός ο διαλόγος και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και να επενδύσουμε σε αυτόν. Και αυτό που αναφέρθηκε στο τέλος ομιλησίας κύριε Βάγνερ θα ήθελα να το υποστηρίξω. Είπατε ότι υπάρχει, χρειαζόμαστε ένα άμεσα ένα ταμείο ε, πολιτιστικό ώστε να μπορέσει να υπάρξει διάλογος, συνομιλίες σε όλες τις ε, χώρες, ε, να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους βάσει ενός κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων βέβαια, αλλά για να τους δώσουμε και περισσότερες ε, ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε αυτό το άνοιγμα, να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε τις διανέξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμετάσχουμε όλοι σε ένα κοινό πολιτισμικό έργο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή ΑΦΕΤ να το λάβει υπόψη να κάνουμε περισσότερα επί του θέματο μέσα στου επόμενου μήνε και τα χρόνια. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Πεστάλτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ του συναδέλφου και την Πρόεδρο την κυρία Κώστα και του συζητητέ και του ομιλητέ για την ποιότητα των ομιλιών του. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Διότι ο συσχετισμός εξωτερικών σχέσεων και πολιτιστικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές παραβλέπεται, παρότι είναι προφανής, διότι ο πολιτισμός είναι ε, ο καλύτερος πρέσβης ε, των αξιών που υπερασπιζόμαστε εμείς. Και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, τόσο δύσκολες εποχές, ε, λόγω της εμφάνισης φονταμεσταλιστών και ριζοσπαστικοποίησης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή στη διενέξη μεταξύ πολιτισμών και αυτή η επίθεση στο Μουσείο Μπάρδο στην Ισία, το οποίο είχα επισκεφθεί, ε, μας λένε κάτι. Δεν είναι τυχαίο που η τρομοκρατία, οι τρομοκρατία χτυπούν πρώτα τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που δεν έχει σύνορα, που εμπλουτίζει αμοιβαία τα διάφορα μέρη, χωρίς ε, να επιβάλλει σχέσεις ισχύω μεταξύ τους. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε συγκεκριμένα έργα και έχετε δίκιο κύριε Βάγνερ όταν μιλάτε για αυτό το άμεσο ταμείο όπως ε, και το πολιτισμικό πρόγραμμα στην Τινησία που θα βοηθήσει τη δημοκρατική μετάβαση που μέχρι τώρα φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα και εκεί μπορεί να βοηθήσει και αυτό το εικονικό μουσείο της Μοσούλης πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απόλυτα αλληλένδετες η πολιτιστική, η πολιτιστική πολιτική και οι εξωτερικές ε, υποθέσεις. Βοηθούν την αξιοπιστία μας και μια δράση δική μας θα αξίζει πολλά περισσότερα από μια πρωτοβουλία ενός μόνο μέλους. Αν παραμείνουμε πιστοί στο σκεπτικό μας ότι υπερασπιζόμαστε την πολυμορφία, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τον πολιτισμό ώστε να ιτηθούν οι δυνάμεις του φανταμεταλισμού από τις δυνάμεις του πολιτισμού. Ευχαριστώ συνάδελφος ο κύριος Πέτρον. Πέτρελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαροποιεί ιδιαίτερα η συζήτηση αυτή σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις συστάσεις και τα μηνύματα κλειδιά συμφωνώ, ο πολιτισμός παρεχτερά στις δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι προς τα εκεί πρέπει να προχωρήσει η πολιτική αναγνωρίζοντας την πολιτιστική ταυτότητα και χρησιμοποιώντας την πολιτιστική ταυτότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ενίοτε αυτός είναι ο καλύτερος, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ εμάς και των υπολείπων. Να προσθέσω επίσης ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτευχθεί μέσα σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν έχουμε ακόμα ενώσει την Ευρώπη. Εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του πολιτισμού. Όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι ανταλλαγές, τόσο πιο πολύ ενοποιημένη θα είναι η Ευρώπη. Και η τρίτη μου παρατήρηση επισκέφθηκα με μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του συναδέλφου μα στην Ινδία. Σε όλα τα επίπεδα οι συνομιλητέ μα τόνισαν ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα στον τομέα του πολιτισμού. Και τέλο, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να διοργανώσει ένα ε, φεστιβάλ κινηματογράφου και είδα με τα ε, μάτια μου πόσο σημαντική ήταν αυτή η εκδήλωση για τους πολίτες μας, για τους κινηματογραφικούς παραγωγούς μας, αλλά και για εμάς. Καταφέραμε να επιτύχουμε ε, τρία πράγματα με μία απλή κίνηση. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό που προωθεί το έργο μας. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps the most exciting debate. initially. είναι η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση και που σε σχέση με μας και για την πολιτική συμμετοχή μετά από την πιστική επίπτωση που είχαν ως καλλιτέχνε, για παράδειγμα με πιλωτικά προγράμματα βλέποντας τις δυνατότητες πώς θα μπορούσαν δημιουργοί, ε, παραγωγή πολιτισμικού έργου να μπορέσουν από όλα, από όλους τους τομείς να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν όσον αφορά ευάλωτα κράτη και καταστάσεις κινδύνου. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω εγώ είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα συνεργάζουν ο ένας δίπλα στον άλλον και θα μαθαίνει ο ένας από τον άλλο. Η δημιουργία νέου ε, καλλιτεχνικού έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση. Και για την διαπολιτισμική Ευρώπη όπου είχα ξεκινήσει και έτσι συνέχισα την πολιτισμική, πολιτική μου δράση θυμάμαι όταν επισκεφθήκαμε τη Βόρεια Ιρλανδία η τέχνη ήταν ένα πολύ σημαντικό μέσο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία ενός ειρηνικού ε, κλίματος ε, ε, πολιτικής και πολιτισμικής ε, συμβίωσης, ε, να δημιουργηθούν γέφυρες, να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας νέος κόσμος όπου οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τις διαφορές τους και θα βρουν τα κοινά στοιχεία που τους ενώνουν ως ανθρώπους και θα υπάρχει δυνατότητα ανάληψης νέων πρωτοβουλειών ώστε να μπορέσουν να, συμβιώσουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Το προηγούμενο καλοκαίρι τον Αύγουστο επισκέφθηκα μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων όπου νέοι Ουκρανοί και νέοι Ρώσοι και νέοι Ρουμάνοι και νέοι Βρετανοί συνομιλούσαν, συνεργαζόντουσαν χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό ως εργαλείο, ως μέσο, ως ένα εργαλείο για να εκφράσουν αυτά που ήταν σημαντικά για αυτούς βρισκόντουσαν σε ένα δωμάτιο αυτοί οι νέοι άνθρωποι ε, και συζητούσαν και συμβίωναν ενώ οι ενήλικες έξω από αυτό το δωμάτιο ο ένας πολεμούσε κατά του άλλου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η συνεισφορά για το μέλλον και την καλωσορίζω θερμά. Edward παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να εκτιμήσω το γεγονός ότι και να το χαιρετήσω ότι με αυτή τη σύνθεση διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από δύο ξεχωριστές κοινοβουλευτικές επιτροπές και για μια πολύ σημαντική συνεισφορά για τα πολιτισμικά θέματα στη συζήτηση αυτή, πράγμα επικοδομητικό. Κάποιες παρατηρήσεις από τη θέση μου ως εισηγητού για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να πω. Είμαι πεισμένος ότι η Ευρώπη έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στο να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτισμική διπλωματία. Ιδιαίτερα όταν έρχεται η ώρα οι χώρες εκείνες που γεωγραφικά βρίσκονται κοντά στην εγκύτητα της Ευρώπης, η πολιτισμική συνεργασία να είναι ένα σημαντικό μέσο και εργαλείο της χείρας που τίνουμε φιλίας προς τους γείτονες μας Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ευδιάκριτος χαρακτήρας της πολιτισμικής αυτής συνιστώσας ως ε, ε, χαρακτηριστικού. Θα πρέπει να υπάρχει διάλογος υψηλού επίπεδου των αρμοδίων για πολιτισμικά θέματα σε σχέση με την ΕΕ. Κάνοντας αυτό μπορούμε να έχουμε θετικές επιπτώσεις σε καταστάσεις όπου θα πρέπει να αναζητηθεί επίλυση σε θέματα σειράξεων και συγκρούσεων και δημιουργίας ειρηνευτικών πρωτοβουλειών και δυνατοτήτων όπως προναφέρθηκε. Έχουμε ήδη κερδίσει αυτά τα βιώματα και αυτή την πείρα από πολλές χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και πρέπει να είμαστε σε θέση και στη γειτονία μας να τα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης υποστήριξη για τις ανταλλαγές ε, πολιτισμικές ε, αλλαγές και, ε, ανταλλαγές και συνεργασίες. Η ανταλλαγή αυτή και σε σχέση με το ανθρώπινο δυνατό δυναμικό είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στις δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς. Και τέλος, λαμβάνουμε υπόψη και θα την λάβω υπόψη στη σύνταξη της πολιτικής γειτονίας όλων αυτών των προτάσεων. Θα τις λάβω υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να προσθέσω τη φωνή μου και να αναφέρω τα δικά μου βιώματα και τη δική μου πείρα. Πριν γίνω Ευρωβουλευτής, αυτό που έκανα ήταν ότι σε σχέση με την ουγγρική ουκρανική πολιτισμική, ας το πω έτσι, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα είχα μελετήσει και κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, όπου η πολιτισμική, πολιτισμική διπλωματία θα μπορεί να χρησιμοποιείται. Τα πολιτισμικά θέματα και ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά είναι μεγάλη σημασίας θα πρέπει να κινήσουμε ότι οι χώρες, τα κράτη έτσι θα εκπροσωπούνται στο εξωτερικό και έτσι με τα διαφορετικά πολιτιστικά ιδρύματα θα πρέπει να δρούμε. Τα πολιτισμικά ιδρύματα της ε, Ουγγαρίας ε, ε, κατά τα τέλη του προηγούμενου αιώνα είχαν δραστηριοποιηθεί σε διάφορες χώρες και είχαν επεκτείνει και είχαν διαδώσει την ουγγρική πολιτισμική κληρονομιά και τα δικά μας χαρακτηριστικά. Και άλλες δραστηριότητες είναι σημαντικές. Αν κάποιος δημιουργός από την καλλιτεχνική σκηνή ή ένας επιστήμονας για παράδειγμα με την ατομική του δράση συνεισφέρει για να υπάρξει συνεννόηση και ε, συναλλαγή είναι πολύ σημαντικό και αν συγκρίνουμε τις δραστηριότητες, για παράδειγμα στα σχολεία, μέσω των ε, δασκάλων, χωρίς ε, τέτοιες, ε, τέτοια θεμέλια και προαπαιτούμενα δεν μπορούμε να έχουμε πολιτισμική δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα έχετε εσείς τον λόγο, παρακαλώ. Μαραγκάλ, ευχαριστώ. Μαραγκάλ, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία. Είχαμε συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για την πολιτισμική κληρονομιά. Φαίνεται φυσικά ότι είναι η θετική συνέχιση όλων αυτών, επικεντρωνόμενη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και παγκόσμια τι μπορεί να γίνει. Μία αυτοκριτική όμως που θα μπορούσαμε να κάναμε στην Ευρώπη να αναφέρω στη διαχείριση των σχέσεών μας με άλλες χώρες νομίζω ότι πάσχουμε από κάτι. Δεν ξέρω αν είναι αφαιρία ή αν είναι ευρωκεντρισμός σαν να είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος θα αφομοιώνει και θα ε, επικεντρώνεται στο δικό μας πολιτισμό και στη δική μας ε, πολιτισμική κληρονομιά. Έτσι δρούμε, αλλά σε πολλές, ε, με πολλές αφορμές ευρισκόμενοι στην Τουρκία για παράδειγμα, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Όμως η γλώσσα μας σε σχέση με την Τουρκία εξακολουθεί να είναι δαιμονευτική πατρο, σαν πάτρονες, σαν να έχουμε το πάνω χέρι και να δίνουμε μαθήματα στους Τούρκους πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε και να μπορούμε να διεκδικούμε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου με τον σωστό τρόπο όμως, με το σεβασμό εναντί των άλλων και όχι με ομό, με, έναν ε, ας το πούμε έτσι ε, σόλικο τρόπο. Αυτό είναι το ε, σημείο επί της ουσίας που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πώς θα μπορούμε να συσχετιστούμε λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό και τις ελευθερίες των άλλων ώστε από κοινέ αξίες να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε κάτι από κοινού. Αυτό ισχύει και για, τα, για τις σχέσεις Ευρώπης με άλλες χώρες, αλλά ισχύει και για την ίδια την Ευρώπη, σε σχέση δηλαδή με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου, των χωρών του Κέντρου ή της Ανατολής και του, της Νότιας Ευρώπης, που είναι, ας το πω έτσι, ε, χαρακτηρίζονται αυτές οι σχέσεις ε, από τέτοιου είδους ε, ας το στάσεις και μια ε, γλώσσα ή ένα τρόπο ε, έκφρασης ε, γλωσσικό που βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να είμαστε πολύ πιο θετικοί και αποτελεσματικοί αν λάβουμε αυτά υπόψη. Ευχαριστούμε κύριε Μαραγκάλη. Και τώρα θα δώσω τον λόγο <clears throat> στον κύριο από τους εκπροσώπους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Απλά και μόνο να πω ότι εμείς ε, από την πλευρά της υπηρεσίας μας ήδη δραστηριοποιούμεθα έντονα στην πολιτισμική διπλωματία και ο συνάδελφος ε, εξεβονίμων και πιο πέρα ακόμα ε, που είχαμε δραστηριοποιηθεί και πριν από 1,5 χρόνο. Εδώ όσον αφορά την εφαρμογή των προπαρασκευαστικών δράσεων και ε, υπό αυτό το πρίσμα που παρουσιάστηκε αναπτύσσουμε δράσεις, αναφέρθηκε η Ουκρανία και προετοιμάζουμε και την ε, δράση όσον αφορά τις ε, άλλες μας πτυχές. Ωστόσο, εντάσσουμε αυτές τις πτυχές στην κανονική μας πολιτισμική δράση, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα σημειωθεί πρόοδος και θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Ποια πρέπει να είναι τα στοιχεία αυτά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσουμε από μια καθαρή πολιτισμική διπλωματία που είναι σημαντική βέβαια να εμπλέξουμε και άλλους δράστες που θα συμμετέχουν. Πολίτες προς πολίτες για παράδειγμα ή τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις και την ε, οικουμενική εμπλοκή και πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα κράτη που συναπαθίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, διεθνείς σχέσεις και στην πολιτισμική διπλωματία. Υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο που είναι η ανάπτυξη ας το πω έτσι, των, της δραστηριοποίησης νέων εμπλεκομένων, του ιδιωτικού τομέα, διαφορετικών τομέων του ιδιωτικού τομέα που θα μπορούν να συμμετέχουν. Και θα αναφέρω και το τελευταίο στοιχείο, το οποίο είναι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ευάλωτος ευαίσθητος χαρακτήρας ε, των ε, πολιτισμικών θεμάτων και ε, όπως και στην Ισία καταδείχθηκε πρέπει κατεπηγόντως να δράσουμε ώστε να υπάρχει δυνατότητα το δυναμικό άμεσης αντίδρασης και ανάληψης πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού τώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σύντομα θα μιλήσω κι εγώ. Πολύ που βρισκόμαστε εδώ σε αυτήν την ε, συζήτηση, όπως είπε και η Σάνα, εδώ και καιρό ασχολούμαστε με το θέμα και συνεργαζόμαστε αυτή την εποχή με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Εξωτερικών ε, Σχέσεων και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε κάποιες από τις συστάσεις προπαρασκευαστική δράση. Πρέπει όμως να πάμε ακόμα πιο μακριά για να έχουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Βάκνερ αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Στακτίν έχει τώρα το λόγο για να σχολιάσει τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών και μετά ο κύριος Βάκνερ και θα ολοκληρώσουμε με την κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας, τα ενδιαφέρον σας, τις παρατηρήσεις σας. Δεν θα σας σχολιάσω τα δικά σας τα σχόλια. Αυτό που θα κάνω είναι ότι θα θέσω ένα ερώτημα. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την πρόταση Βάγνερ όσον αφορά τον πολιτιστικό μηχανισμό της προπαρασκευαστικής δράσης. Ρωτώ λοιπόν, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μια τέτοια πρόταση. Όλοι θέλουμε συγκεκριμένες δράσεις. Πολλά γίνονται. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν κάποια βήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα, οπότε είναι καλή, σωστή στιγμή τώρα να περάσουμε σε πιο συγκεκριμένη δράση και όλες αυτές τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες να τις δούμε στην πράξη στο μέλλον. Άρα ερώτηση βασικά έχω, όχι σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε. Κύριε Βάγκνερ, η σειρά σα. Και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έχουν ήδη γίνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα στα τέλη του θέλει να έχει ιδρύματα Κομφούκη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Αυτό βέβαια δείχνει την αναγκαιότητα για μακρόχρονη στρατηγική. Χαίρομαι πολύ πάντως για τις θετικές αντιδράσεις σας. Χρειαζόμαστε όμως κάποια μέσα, κάποια εργαλεία που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ γρήγορα. Ο πολιτισμός δεν απαιτεί τεράστια ποσά, ούτε περίπλοκη τεχνολογία. Χρειάζεται ανθρώπους. Όταν μιλάμε με τους νέους σήμερα, και είμαι εγώ αρκετά μεγάλο, οπότε μπορώ να μιλήσω για νέου. βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον του για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέση με το θετικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνεί υποθέσει. Ο πολιτισμό λοιπόν είναι ένα από του τομεί στον οποίο θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιείται. Αυτό είναι που λένε, Του βοηθάει να επικοινωνήσουν και μεταξύ του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα. Πρόεδρο ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάγκνερ. Χαίρομαι για τον ενθουσιασμό που διαπίστωσα στη συζήτησή μας και από τους ευρωβουλευτές που παραμένουν στην αίθουσα και που δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στην συνεργασία όλων μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους εμπειρογνώμονες, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο ένα πολιτικό σχέδιο, είναι και ένα πολιτισμικό, πολυπολιτισμικό θα έλεγα ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ειρήνης, στην καλύτερη κατανόηση στα πλαίσια των κρίσεων που συναντάμε γύρω μας. Είναι πολύ θετικά λοιπόν όσα ακούσαμε σήμερα. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την κυρία Κώστα να καταλήξει στα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι αυτή εδώ αποτέλεσε την πρώτη σημαντική ευκαιρία, το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδρομή που εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να συνεργαστούμε επί ενός θεμάτος που μου φαίνεται κατεπήγον αφενός, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Επίσης όμως και για να ενισχύσουμε μια στρατηγική που θα αξιοποιήσει τον πολιτισμό, όπω προέκυψε από τη συζήτηση εδώ, θα αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό ως ένα παράγοντα που θα επηρεάσει σημαντικά την εξωτερική μας πολιτική. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των ακραίων θρησκευτικών πολιτιστικών θέσεων που ε, δεν επιτρέπουν το διάλογο και να δώσουμε εμείς μια απάντηση σε αυτό, μια απάντηση προηγμένη να υπενθυμίσουμε ότι φέτος κλείνουν 10 χρόνια τη συνθήκη της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία και εμείς στην Επιτροπή μας έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε μια ακρόαση που θα λάβει χώρα μέσα στους επόμενους μήνες ε, και που θα αφορά την πολιτιστική πολυμορφία και την πρόθεση του πολυ... πολιτισμικού διαλόγου επισκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια ακρόαση για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στον πολιτισμό. Εάν ενώσουμε, πιστεύω, τις δυνάμεις μας, ε, οι δύο επιτροπές ΑΦΕΤ και πολιτισμού και ε, αναλάβουμε στεναρή δράση προσαρμόζοντας ε, τη δράση της κάθε επιτροπής και ξέρω ότι έχει δεσμευτεί και η κυρία Μογκερίνη, είπατε εκπρόσωπος, Σήμερα μιλήσαμε και για δύο ανθρώπους που είναι σύμβολοι για αυτό ακριβώς το θέμα της κυρίας Μογκερίνη. Εγώ λοιπόν θα συζητήσω με τους συντονιστές της Επιτροπής μου και ελπίζω να κάνετε το ίδιο και στη δική της Επιτροπή ώστε να δούμε ε, ποια θα μπορούσε να είναι η πρωτοβουλία, αν θα μπορούσε να είναι κοινή. Πιστεύω θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε κάνει μια σχετική παρέμβαση, αλλά μια τέτοια κοινή αποφασιστική δράση δική μας ε, πιστεύω θα ήταν πολύ δυνατή. Σύμφωνα με πολλές από τις προτάσεις που ακούσαμε, συνεργάζομαι και με τον κύριο Διακόνου για το θέμα αυτό τη σημαντική αυτή έκθεση για την πολιτιστική κληρονομιά προβλέπεται για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής για την εξωτερική δηλαδή διάσταση της ε, προστασίας, ε, της πρόληψης, της καταστροφής ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σημαντικό κομμάτι και αυτή η έκθεση αλλά πρέπει να μελετήσουμε και τους πέντε τομείς που αναφέρατε κύριε Βάγκνερ το ταμείο που ανέφερε και ο συνάδελφος του Μήπως αυτό όμως ενταστεί στις αρμοδιότητες της ΑΦΕΤ περισσότερο, διότι εντός των εξωτερικών δράσεων το θέμα αυτό του να δούμε κατά πόσο μπορεί να επεξεί κάποιο ταμείο ειδικά για την πολιτική, εξωτερική πολιτική εντός του οποίου θα υπάρχουν διμερείς ε, συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Μιλήσαμε για μια εμπειρογνωμοσύνη που έχει ήδη η Ευρώπη περισσότερο στο μέτωπο των Βαλκανίων όπω είπαμε πριν, αλλά αυτή τη στιγμή στρατηγική προτεραιότητα άμεση αποτελούν οι χώρε γύρω από τη Μεσόγειο. Και είμαι βέβαιη ότι όπω συνέβαινε ανέκαθεν, επειδή έχουμε συνείδηση το ότι μα συμφέρει μια ισχυρή συνεργασία για την πολιτική κληρονομιά, αλλά και στο πλαίσιο των σχέσεων και στον τομέα τη δημιουργικότητα ε, στον κινηματογράφο, ε, Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα θέση της Ευρώπης ενώπιον των χωρών της Αφρικής, της Μεσογείου που κατά κάποιο τρόπο έχουν ανατρακτεί τα τελευταία χρόνια από κάποιες ε, λάθος ε, παρανοήσεις. Ε, Ένα άλλο ζήτημα που θεωρώ είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα είναι οι δυνατότητες πρόληψης και διαχείρισης διενέξεων δύσκολα θέματα. Εδώ αναφέρομαι σε αυτά που αναφέρουμε ως soft skills και ε, επίσης ε, μην ξεχνάμε την αμοιβαιότητα σε αυτή τη νέα εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου προβλέπεται αυτή η μη κυδαιμονευτική μορφή ε, συνεργασίας και αμοιβία συνεργασίας. Αυτό πιστεύω θα ενίσχυε ιδιαίτερα την κοινωνία των πολιτών και όλους τους νέους που μέσα σε αυτή την πραγματικότητα σίγουρα θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα για τέτοιε σχέσει. Εμεί έχουμε κάποιε εμπειρίε όσον αφορά και το πρόγραμμά μα Creative Europe, να δώσω μόνο αυτό το παράδειγμα, όπου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στι διεθνεί σχέσει, όχι μόνο εντό των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των χωρών τη ε, ε, γειτονίας μας. Αυτά τα δίκτυα πολύ συχνά φέρνουν εκπληκτικά αποτελέσματα, φέρνουν κοντά ανθρώπου, κινητοποιούν ανθρώπου Και στο πλαίσιο του Horizon, όπω είπαμε πριν, ε, μπορούμε να προσδιορίσουμε ε, κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες που όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία για την ανακαίνιση μνημείων, αλλά και πρωτοβουλίες που σχετίζονται περισσότερο με ανθρώπους ε, και δίκτυα. Κατά την άποψή μου λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε ως εξή. Εγώ θα φροντίσω να συζητήσω με τους συντονιστές ε, της Επιτροπής Πολιτισμού για να προσδιορίσουμε το επόμενο βήμα κοινοποιώντας το σε εσά, ε, εφόσον συνεργαστούμε ενεργά και σε περίπτωση μια τέτοια συνεργασία πιστεύω τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας και για αυτή την ισχυρή σα βούληση που είναι και δική μας βούληση για μια ορατή στρατηγική αναγκαία αυτή την εποχή. Ευχαριστώ κύριε Κώστα, ευχαριστούμε τους εμπειρογνωμονές μας, ευχαριστώ όλους ε, που Μείνατε εδώ μέχρι τις 6.45. Ευχαριστούμε και τους Δερμήνης. Έχει κλείσει η συνεδρίαση. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα το απόγευμα στην Επιτροπή Άρθρα. Ευχαριστούμε.